και κύριοι, η Ραζάμ Ζάιτσουνου ε, τιμηθήσαμε το βραβείο Ζαχάροφ πριν από δύο μήνες απήχθη μαζί με το σύζυγό της και ακόμη έναν ε, ε, αγωνιστή για τα ανθρώπινα δικαιώματα από μια ομάδα έξω από τη Δαμασκό δεν είναι γνωστό το που βρίσκεται. Τους τελευταίους δύο μήνες δεν έχουμε καμία είδηση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί τη ε, απευθύνει έκκληση για την ταχύτατη απελευθέρωση της κυρίας Ζαϊτσουνή. Πρόκειται για έναν άνθρωπο που αγωνίστηκε και αφιέρωσε τη ζωή του στα ανθρώπινα δικαιώματα και την ελευθερία. Έχει αντιμετωπίσει απειλές τόσο από το καθεστώς Συρίας όσο και από τις ομάδες των αντικαθεστωτικών αλλά δεν είναι και η μόνη η οποία έχει απαχθεί, βασανιστεί, κρατηθεί παράνομα. Είναι ένα ακόμα από τα θύματα των, του πολέμου αυτού. Πολλές φορές στη Συρία χρησιμοποιείται προκειμένου να καταπιεστεί περαιτέρω ο λαός, η κοινωνία της Συρίας ε, ως όπλο ο βιασμός. Πρέπει να τον καταδικάσουμε με κάθε τρόπο και πριν από δύο μέρες ξεκίνησε η σύνοδος για το θέμα αυτό. Πρέπει να τοποθετηθούμε, να υποστηρίξουμε άτομα και οργανώσεις που προστατεύουν και προσφέρουν βοήθεια στις γυναίκες που έχουν πέσει θύματα βιασμού ώστε να μπορούν να ξαναγυρίσουν σε μια ομαλότητα στη ζωή τους, αλλά ταυτόχρονα και να καταγράψουν και να τεκμηριώσουν τα εγκλήματα αυτά που διαπράττονται. Για άλλη μια φορά απευθύνουμε έκκληση για την απελευθέρωση της τιμηθής σας με το βραβείο Ζαχάροφ, Ρεσάζα και στις ανακοινώσεις. Η κυρία Φραντσέσκα Μπαρατσού από τις 28 Φεβρουαρίου έχει αναλάβει καθήκοντα στην Ιταλική κυβέρνηση. κυβέρνηση. Ο κύριος Κλάους Χάινερ Λένε από 1 Μαρτίου 2014 ε, αναλαμβάνει καθήκοντα ως